Πριν να κηρύξω την έναρξη τη Συνόδου Ολομέλεια, ήθελα να εκφράσω εξ ονόματο του Κοινοβουλίου τα θερμά μα συλληπιτήρια προ τα τις οικογένειες των θυμάτων των πρόσφατων θρησκευτικών ε, διώξεων και τρομοκρατικών επιθέσεων. Η γενοκτονία των χριστιανών δεν έχει πάψει.